2012 διεκόπη συνεχίζεται με σημερινή ολομέλεια. Τα πρακτικά και τα εγκεκριμένα κείμενα της Συνόδου της 13ης 12ου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, αντιρρήσεις. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι,